Κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε τη συνεδρίαση. Θα ήθελα να σας ανακοινώσω ορισμένε αλλαγές στην ημερήσια διάταξη. Σας έχουν ήδη σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδραμείο για τη σημερινή συνάντηση τα σημεία 4 και 5 έκθεση Γέλκο Κασίν για τη Σερβία και το 5 επίσης, δεν θα συζητηθεί το θέμα αυτό γιατί ο κακός καιρός τον έχει αποκλείσει τον κύριο Κατσίν και θα είναι στις Βρυξέλλες αύριο και θα ψηφίσουμε την έκθεσή του. Η ψηφοφορία προβλέπεται όπως το λέγει η ημερήσια διάταξη στις 4.30 αύριο. Κύριε Τάνοκ, ε, εισηγητής για το Μαυροβούνιο, συμφώνησε ο κύριος Τάνοκ και τον ευχαριστούμε γι' αυτό έτσι ώστε να συζητήσουμε το θέμα του για τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Μαυροβουνίου σήμερα σαν πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Τα υπόλοιπα θέματα της σημερινή συνεδρίασης θα ε, διεξαχθούν κανονικά. Πρέπει να γνωρίζετε όμω ότι η συζήτηση για τις διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκή Ένωση Λιβύη ε, ίσως να συζητηθεί λίγο νωρίτερα σχετικά τώρα με την αυριανή συνεδρίαση της ε, Τετάρτης 1ης Δεκεμβρίου. Μετά από τα γεγονότα τα οποία διαξήχθησαν στις 8 Νοεμβρίου στο στρατόπεδο Τακταϊνιζίτ ε, και μετά από τις πάρα πολλές αντιδράσεις που ε, συνέλεξαν οι συντονιστές, ο πρόεδρος Αλμπερτίνη αποφάσισε να εγγραφεί το θέμα αυτό στην αυριανή ημερήσια διάταξη. Έχουν σταλεί ε, ε, προσκλήσεις στον Μαροκινό Υπουργό Εξωτερικών και στον κύριο Μωάμεντ Σάλαμους Νταλέκ εκπρόσωπο του μετόπου Πολυσάριο υπεύθυνο για τις εξωτερικές σχέσεις όπως και προς τον κύριο Μοχάντ Μπελενζή, Υπουργό Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Αλγερίας, για να υπάρξει μια κοινή συζήτηση μαζί τους. Η απουσία απαντήσεων από πλευράς της Αλγερίας αποφασίστηκε να περάσουμε σε δύο και χωρισμένες ανταλλαγές απόψεων. Η πρώτη θα γίνει αύριο από τις 9 και 4 μέχρι τις 10 το πρωί την παρουσία του κυρίου Ουντ Σαλέκ εκπροσώπου του μετόπου Πολυσάριο και η δεύτερη ανταλλαγή απόψεων αύριο από τις 11 μέχρι τις 11 και 45 τη παρουσία του κυρίου Φασί Φέρι, ο οποίος είναι υπουργό Εξωτερικός του Βασιλείου του Μαρόκου. Το σημείο 9 ε, για την Κροατία, μουσείο δηλαδή του κυρίου ε, Σβόμποντα, ε, στις 11.45 αύριο. Τώρα για τη δεύτερη συνεδρίαση της Πέμπτης, ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Πίτερ Φέις, ειδικό εκπρόσωπο στο κοσυφοπέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 10.30 και όχι στις 11.15. Θα ακολουθηθεί από την έκθεση της κυρίας Μακοβέη υπεύθυνη τη ομάδα εκλογική παρατήρηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τι εκλογέ οι οποίε διεξήχθησαν στη Μολδαβία την προηγούμενη Κυριακή. Αυτά δεν ξέρω αν υπάρχουν αντιρρήσεις γύρω από την ημερήσια αυτή διάταξη και τι αλλαγέ που προτάθηκαν. Δεν φαίνεται να υπάρχουν αντιρρήσεις και σα ευχαριστώ γι' αυτό. Θα υποβάλω τώρα προς έγκριση τα πρακτικά της συνεδριάσεώς μα της 14ης Οκτωβρίου δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, συνεπώς θεωρούνται δεκτά τα πρακτικά. Μια ανακοίνωση της Προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ασφάλεια στην Κορεατική Χερσόνησο και γενικά στην Ανατολική Ασία. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Η Επιτροπή μας θα εξετάσει, είναι αυτονόητο, από κοντά την ε, εξέλιξη των διπλωματικών πρωτοβουλειών που έχουν ξεκινήσει ήδη και στα πλαίσια της ομάδας των έξι, των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε έξι και δεν εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τις πρωτοβουλίες που μπορεί να ληφθούν στα πλαίσια του Συμβουλίου Ασφαλείας. Άμεσα όμως θα ήθελα να ενημερώσω τους ενδιαφερομένους συναδέλφους ότι η αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κορέα ξεκινά αυτή τη στιγμή μια συνεδρίαση η οποία είχε προγραμματιστεί εδώ και αρκετό καιρό αλλά παίρνει διαφορετική σημασία λόγω της συγκυρίας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αυτής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα περιγράψει την πολιτική κατάσταση, την κατάσταση στον τομέα ασφαλείας και τα προβλήματα τα ανθρωπιστικά και προβλήματα διατροφής που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός της Βόρειας Κορέας. Πρώτο σημείο λοιπόν της ημερήσιας διάταξης είναι πλέον η έκθεση του κυρίου Τάνοκ για την υποψηφιότητα του Μαυροβουνίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με πολύ μεγάλη χαρά παρουσιάζω την πρώτη πρόταση της έκθεσής μου μετά από τις πρόσφατες συστάσεις τις οποίες έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το Μαυροβούνιο έτσι ώστε να δώσουμε στη δημοκρατία του Μαυροβουνίου την ιδιότητα του υποψηφίου μέλους, αν και δεν συστήνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσουν άμεσα οι διαπραγματεύσεις, αλλά υπάρχουν διάφορα επίπεδα, τα οποία στάδια, στα οποία πρέπει να φτάσει η χώρα αυτή, πριν ξεκινήσουμε επίσημα την συζήτηση των κεφαλαίων του κοινοτικού κεκτημένου. Στην έκθεσή μου τα αναφέρω όλα αυτά λέγοντας ότι αυτό το μοντέλο, το πρότυπο το οποίο όλον και περισσότερο υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσυνδέει δηλαδή την ιδιότητα του υποψηφίου μέλους με την έναρξη των διαπραγματεύσεων από την άλλη ε, μου δημιουργεί αρνητικές σκέψεις θα έλεγα. Αυτό το έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την Μακεδονία λέει ο μιλητής το ίδιο κάνει τώρα και με το Μαυροβούνιο. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για ένα κεφάλαιο, τουλάχιστον για τη μεταφορά νομοθεσία από το κοινοτικό κεκτημένο στην εσωτερική νομοθετική τάξη τη υποψήφια χώρα και το κλείσιμο του συγκεκριμένου κεφαλαίου που αφορά την εφαρμογή των συγκεκριμένων αυτών διατάξεων και όλων των υπολείπων δυνατοτήτων που υπάρχουν για την αύξηση πίεσης, μεγαλύτερης πίεσης Πρόκειται για νέα, νέα σενάρια θα έλεγα. Νομίζω ότι η Επιτροπή μας, αυτή εδώ η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο δεν μπορούν παρά να δεχτούν Βέβαια λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η αποσύζευξη δεν θα πρέπει να καταστεί αθέμητη, δεν θα πρέπει να είναι μακροπρόχρονη και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να φέρει σε αδράνεια όλες τις προσπάθειες της χώρας να έρθουν κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανεξαρτήτως ουσίας. Όπως αναφερθήκαμε ήδη το Μαυροβούνιο και το είχε πει ο αρμόδιος επίτροπος για την διεύρυνση, είναι καλά νέα. Είναι μια νέα χώρα, νεοπαγής χώρα, μικρή χώρα. Υπάρχουν 24 παράγραφοι που εξηγούνται όλα αυτά τα θετικά λοιπόν. Αυτό βέβαια δεν αντικατοπτρίζει, αυτά δεν αντικατοπτρίζουν το μέγεθος της χώρας, αλλά λόγω του ότι έχουμε να κάνουμε με θετικά θα έλεγα αρκετά. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα παρά θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεσή μου, θέματα δηλαδή κράτους δικαίου, και θέματα αύξησης της προσπάθειας καταπολέμησης της διαφθοράς και του εγκληματική δραστηριότητας. Δεν έχουμε τα προβλήματα που έχουμε με άλλες χώρες όπως η Αλβανία που δεν είναι πλέον υποψήφια χώρα λόγω της ε, κοινοβουλευτικής παράλυσης που την χαρακτηρίζει. Το Μαυροβούνιο είναι μια λειτουργούσα δημοκρατία, είναι μια σταθερή οικονομία, έχει de facto υιοθετήσει το ευρώ σαν ε, μέσο ανταλλακτικό την χάνει των διευκολύσεων στον τομέα των θεωρήσεων, δεν χαρακτηρίζεται από μασικές ε, μετακινήσεις πληθυσμού ή από καταχρήσεις των συμφωνιών Σέγγεν, δεν υπάρχουν πολλά προβλήματα ε, μεθοριακά ε, με τις γειτονικές χώρες, εκτός από ένα μικρό πρόβλημα με την Κροατία, το οποίο θα μπορέσουμε να το επιλύσουμε και μέσω του παραδείγματος που έθεσε η ρύθμιση του προβλήματος ανάμεσα στην Κροατία και στη Σλοβενία ε, και θα λυθεί το θέμα είτε μέσω ε, δημοψηφίσματος είτε μέσω προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο έχει κάποιες μειονότητες, υπάρχει ένα θέμα με Ρωμά από το Κωσυφοπαίδιο σε ένα συγκεκριμένο στρατόπεδο και τίθεται ένα θέμα για το καθεστώς τους και τις συνθήκες κατά από τις οποίες διαβιούν, αλλά ο αριθμός τους είναι πολύ χαμηλότερος από τις στις γειτονικές χώρες. Υπάρχουν επίσης ορισμένα προβλήματα τα οποία θα πρέπει να ανταποτεπιστούν σε σχέση ε, με τα αντιτιθέμενα οικονομικά συμφέροντα και προσωπικά συμφέροντα των μελών του Κοινοβουλίου και άλλων μελών της εκτελεκτικής εξουσίας ε, για το κατά πόσον θα πρέπει να επιτρέπεται να πληρώνονται ας πούμε από δημόσιες υπηρεσίες αλλά και να έχουν ξεχωριστά ιδιωτικά συμφέροντα. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να δούμε. Υπάρχουν συνεχείς καταγγελίες επίσης ε, λόγω ακριβώς της ύπαρξης του ευρώ εκπλήνσης βρώμικου χρήματος. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά Υπάρχει επίσης μια υποεκπροσώπηση των γυναικών στην δημόσια ζωή αν συγκρίνουμε με τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ είμαι βέβαιος ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ικανοτάτων γυναικών στη χώρα αυτή που μπορεί να φέρει εις πέρας πολλές αποστολές. Υπάρχουν επίσης και κάποιες δύο μικρές κοινότητες ε, ε, γύφτων, όπως επίσης και ασκαλή μιας άλλης ομάδας Ρωμά, οι οποίοι ε, θα προτιμούσαν από ό,τι λέγουν να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσής τους. Πρόκειται λοιπόν για μια μικρή χώρα, έχει κάποιες περιορισμένες διοικητικές ικανότητες η μηχανή δημόσια της χώρας αυτής, και γι' αυτό η, συμπερίληψη της χώρας αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ίσως λίγο πιο θα έλεγα δύσκολη από ό,τι μεγαλύτερες χώρες, αλλά έχουμε παραδείγματα όπως η Εστονία, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα. Νομίζω ότι το Μαυροβούνιο βοηθήθηκε επίσης πολύ και από τη γενεοδορία την Κροατική, που η οποία ήδη μετέφρασε 800.000 περίπου του κοινοτικού κεκτημένου όχι στην ίδια γλώσσα, γιατί αυτό θα προκαλέσει τις αντιδράσεις πολλών, αλλά σε μια γλώσσα η οποία είναι αμοιβαίως κατανοητή από πολλές χώρες. Το Μαυροβούνιο επίσης αυτοπροσδιορίζεται ως οικολογική χώρα, κάτι το οποίο είναι περίεργο για μια χώρα. Έχει πραγματικά εξαιρετικά εντυπωσιακά τοπία και αυτό είναι πολύ θετικό και ιδιαίτερα η πλέον πράσινη των συναδέλφων σε αυτή την Επιτροπή και είναι μια χώρα η οποία πρέπει να αποδείξει βέβαια τι εννοεί ότι είναι πράσινη σχετικά με την προστασία της εθνικής κληρονομιάς. Σε επίπεδο οικονομικό ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι ότι είναι ο μονοκαλλιεργητική. Δεν έχει πάρα πολλέ βιομηχανικές επενδύσεις εκτός από ένα πάρα πολύ μεγάλο χιτήριο το οποίο θα πρέπει τα ταχύτατα να εξυγχρονιστεί. Έχει επίσης τεράστιες ε, ε, δυνατότητες σχετικά με εξαγωγή ηλεκτρισμού και ίσως να δημιουργηθεί και ένα δίκτυο με την Ιταλία το οποίο θα επιτρέπει την εξαγωγή ηλεκτρισμού σε χώρες όπως η Ιταλία οι οποίες πεινούν για ηλεκτρισμό. Αυτό ε, προμηνύει πολλά καλά αλλά κυρίως εξαρτάται από τον τουρισμό η οικονομία της χώρας ο οποίος κυμαίνεται ανάλογα και με το ύψος του ευρώ και με τη γενικότερη πολιτική συγκυρία. Υπάρχει όμως και εδώ όπως και στην ενέργεια πολύ καλή προοπτική. Έχει πολύ καλές σχέσεις με όλες τις χώρες, έχει πολύ καλές σχέσεις και με το Βελιγράδι, όπου τα πράγματα ήταν λίγο ψυχρά στην αρχή, μετά από τον αρχικό αποχωρισμό θα έλεγα, υπήρξαν κάποια προβλήματα της αναγνώρισης του Κωσυφοπεδίου από το Μαυροβούνιο, αλλά οι σχέσεις τώρα είναι καλές ανάμεσα στη Σερβία και το Μαυροβούνιο και νομίζω πρέπει να αναγνωρίσουμε στο Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου ότι έχουν αναγνωρίσει τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων. λέω ο και πράγματι εξέδωσαν ένα ψήφισμα πολύ σημαντικό σχετικά με τη Σρεμπρένιτσα. Νομίζω λοιπόν ότι είπα τα περισσότερα, τα υπόλοιπα περιλαμβάνονται στη γραπτή πρόταση και περιμένω με ενδιαφέρον να ακούσω αυτά τα οποία θα πούν οι συνάδελφοι και τις πιθανές τροπολογίες οι οποίες σίγουρα θα συνεισφέρουν στο να εμπλουτίσουν την έκθεση. Γενικότερα το Μαυροβούνιο νομίζω ότι θα είναι μία από τις ευκολότερα ε, θα έλεγα απορροφήσιμε σε εισαγωγικά χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στην περιοχή της Δυτικής Βαλκανικής. Σας ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Euh, το λόγο κύριος Ντανζό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Τάνοκ για την έκθεσή του. Μας κάνει μια σωστή αποτίμηση της πραγματικότητας, διαπιστώνει επίσης πολύ σωστά πρόοδο, μας απαρίθμησε τα θετικά σημεία αυτής της υποψηφιότητας, χωρίς να αγνοεί όμως και τις αδυναμίες αυτής της χώρας και την πρόοδο που απομένει να επιτελέσει. θα πρέπει να είναι υπερβολικά επίκης και συγκαταβατική η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να είναι πολύ απαιτητική στην πρόοδο. Ε, ιδιαίτερα στο θέμα της δικαιοσύνης και της ελευθερίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι όταν μιλούμε για το Μαυροβούνιο θα πρέπει να κρατούμε τη μνήμη μας ε, ζωντανή, γιατί ήταν κοντά μας σε κρίσιμες στιγμές ευρωπαϊκής ιστορίας και στη σύγκρουση στο Κωσυφοπαίδιο και σε, διάφορες, σε διάφορα διεθνή προβλήματα ευθυγραμμίστηκε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υιοθέτησε απόψεις πολύ κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι μπορούμε κάλλιστα να, έχουμε, και ε, ε, έδειξε ότι μπορεί κάλλιστα να έχει καλές, θέσεις, καλές σχέσεις γειτονίας ε, με χώρες στην οποία ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση όπως η Κροατία και είναι από τις πιο πολυεθνοτικές χώρες των Βαλκανίων. Μόνο το 40% του πληθυσμού των Μαυροβούνιων χαρακτηρίζονται ως Μαυροβουνίτες. Δηλαδή ούτε καν η πλειοψηφία. Είναι πολυεθνωτική αυτή η χώρα. Και εξαιτία ακριβώς τι ευπάθειε που αντιμετωπίζει ο πολυεθνικό χαρακτήρα σε πολλέ χώρε είδαμε ότι στο Μαυροβούνιο δεν υπήρξαν ανοιχτέ πληγέ ή σοβαρέ κρίσει λόγω αυτής της πολυμορφίας. Επίσης, ε, μερικές φορές ε, στυλιτεύουμε δύο χώρε ε, ω συμβολικέ για λόγου διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματο. Όλο τυχαίω, οι δύο αυτέ χώρε είναι το Μαυροβούνιο και Παρ' όλα αυτά, δωροδοκία, αδιαφάνεια, προβλήματα ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη σίγουρα υπάρχουν, μα το επισήμανε και ο εισηγητή. Αλλά αυτό ισχύει για όλε τι βαλκανικέ χώρε, χωρί καμία εξαίρεση. Από τι πιο προηγμένε όπω είναι η Κροατία, ω τι λιγότερο προηγμένε όπω το Κωσυφοπέδιο. Το να τι ε, συνέχεια και να κατονομάζουμε δύο μόνο χώρε δεν νομίζω ότι είναι μια σωστή αποτίμηση τη πραγματικότητα στην περιφέρεια ό,τι αφορά το έγκλημα ή την ε, έλλειψη ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Από αυτή την άποψη η έκθεση του κυρίου Τάνοκ ε, σε πολύ επίκαιρη στιγμή και πολύ εύστοχα μας υπενθυμίζει με αντικειμενικότητα την κατάσταση στο Μαυροβούνιο και συμφωνώ απόλυτα με τους προσανατολισμούς της έκθεσής του. Ε, Ο κύριος Κυρίλοφ. Όχι, κύριε Κορνέλισεν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Τάνο και την έκθεσή του, γιατί πραγματικά ασχολείται με πολλά θέματα που και για μας είναι σημαντικά. Το Μαυροβούνιο, όπως είπατε, είναι μια πολύ μικρή χώρα. Το θετικό αυτής της έκθεσης είναι ότι είναι όλοι γνωστοί μεταξύ τους. Όλοι γνωρίζουν τα πάντα, τους πάντες. Κάτι που κάνει τη χώρα λίγο αντιδραστική στις μεταρρυθμίσεις. Για παράδειγμα, συζήτησα δικαιώματα ομοφιλοφίλων με υπουργού και κοινοβουλευτικούς. Και το πρώτο πράγμα που ρώτησαν τους δερμηνείς ήταν αν πραγματικά είπαν τη λέξη γκέι και άρχισαν να χασκογελάν. Έχει μακρύ δρόμο να διανύσει δηλαδή αυτή η χώρα ε, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των μειονοτήτων, των σεξουαλικών μειονοτήτων, τα δικαιώματα των γυναικών κτλ. Επίσης η χώρα αυτή είναι κάπως αντιδραστική σε ό,τι αφορά την πάταξη της διαφθοράς. Άκουσα πρόσφατες εκθέσει μη κυβερνητικών οργανώσεων που κατήγγυλαν παρενοχλήσεις και μάλιστα ε, κατήγγυλαν ότι τους παρακολουθούσαν μυστικοί πράκτορες. Το Μαυροβούνιο εξαιτία των μικρών διαστάσεών του έχει και κάποια πλεονεκτήματα. Ε, δηλαδή, όσο μικρότερη μια χώρα, ίσως τόσο μικρότερα προβλήματα έχει και τα ίδια προβλήματα σε μεγαλύτερη διάσταση ήταν πιο σοβαρά. είναι μία από τις χώρες που δεν έχει υποστεί από τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες όπως η Ολλανδία για τα θέματα, για τα θέματα της απελευθέρωσης των θεωρήσεων, γιατί σίγουρα δεν έχουμε μαζικές μεταναστευτικές ροές από το Μαυροβούνιο, κατοίκους που να κατέκλυσαν ε, τις ευρωπαϊκές χώρες. Σε ό,τι αφορά το θέμα της απελευθέρωσης των θεωρήσεων, κάτι που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στην έκθεση είναι το πώς ε, χειρίζεται το θέμα της ηθαγένειας στο Μαυροβούνιο. Για παράδειγμα, έχουν μια πρακτική της απόδοσης ε, τιμητικής ηθαγένειας, κάτι που αναπόκειται στη διακριτική ευχαίρεια της κυβέρνησης και δίνουν αυτό το, αυτή την τιμητική θαγένεια σε όποιον ε, κρίνουν ε, ότι τους ε, ικανοποιεί. Οποιοςδήποτε επενδύει μισό εκατομμύριο ευρώ στη χώρα μπορεί να λάβει τιμητική θαγένεια, να γίνει επίτιμος μαυροβουνίτης. Επίσης το γεγονός ότι δεν προβαίνει σε απελάσεις το, Μαυροβούνιο ή δεν εκδίδει μάλλον, δεν προβαίνει σε εκδόσεις είναι κάπως ύποπτο γιατί μπορεί να γίνει ασφαλές λιμάνι και καταφύγιο για εγκληματίες. Ναι, συμφωνώ με τον κύριο Τάνοκ. Είναι θαρρυντικό το γεγονός ότι αυτό αποκαλείται το Μαυροβούνιο ως οικολογικό κράτος, αλλά βλέπουμε τι υφίσταται το περιβάλλον από την ανάπτυξη του τουρισμού. Γι' αυτό και πραγματικά θα ήταν κρίμα να καταστραφεί ο φυσικός πλούτος αυτός, αυτής της χώρας, όχι εξαιτίας εγγενούς αξίας που έχει ο φυσικός πλούτος, αλλά γιατί μία ε, απίχνωση του φυσικού πλούτου θα οδηγήσει σε μείωση και της ε, τουριστικής κίνησης, γιατί οι τουρίστες ε, για το φυσικό πλούτο πηγαίνουν κυρίως στο Μαυροβούνιο. Οπότε οι νέες εξελίξεις όπως εργοστάσια υδροελεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να συνοδευτούν από μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και από προσπάθεια προστασίας και διαφύλαξης του περιβάλλοντος. Θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες για τα θέματα που σας ανέφερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βάγκελ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από ό,τι φαίνεται, στο Μαυροβούνιο είναι αδύνατο να, πούμε κάτι για τη χώρα αυτή και οποιοδήποτε να μιλήσει για τη χώρα αυτή χωρίς να εκδηλώσει τη συμπαθιά του. Γιατί όντως το Μαυροβούνιο είναι μια μικρή χώρα που χρήζει κατανόησης, μεγάλης κατανόησης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι και λόγος ε, αποφυγής οποιασδήποτε κριτικής εις βάρος του Μαυροβουνίου. Γιατί το Μαυροβούνιο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως υποψήφια για ένταξη χώρα. Ο κύριος Στάνο, κατά τη γνώμη μου, στην γνωμοδότησή του, πολύ εύστοχα και ρητά απαρίθμησε στην, ε, στο έργο του, στο πόνημά του και τις θετικές πλευρές, πλευρές αλλά και τις αρνητικές πλευρές της κατάστασης ε, που επικρατεί στο Μαυροβούνιο. Βέβαια παραμένουν εκκρέμει κάποια θέματα. Το Μαυροβούνιο θα πρέπει να τα αντιμετωπίσει στο εγγύς Θα πρέπει για παράδειγμα να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα γιατί θα εξακολουθεί να υφίσταται στο στενό έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρθηκαν θέματα διαφθοράς, κράτους δικαίου, οργανωμένου εγκλήματος, πρόβλημα με την ε, ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Όλα αυτά τα θέματα είναι παρόντα και όλα αυτά τα προβλήματα ταλανίζουν όλες τις ε, χώρες που βρίσκονται σε μεταβατική φάση. Δεν είναι χαρακτηριστικά μόνο του Μαυροβουνίου αλλά σε ορισμένε περιπτώσει είναι πιο εύκολο να εντοπιστούν, να διαγνωστούν. Και όσο πιο μικρή μια χώρα, τόσο πιο καθαρά φαίνονται αυτά τα προβλήματα. Όταν μιλούμε για την ελευθερία έκφραση και την ελευθερία των μέσων μαζική ενημέρωση, είναι προφανέ, είναι ηλιοφανότερο μάλλον, ότι όταν ανακύπτουν προβλήματα, τραβούν αμέσω την ε, προσοχή των διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οι νομοθετικές αρχές του Μαυροβουνίου θα πρέπει να δείξουν μεγαλύτερο βαθμό ευαισθησίας ό,τι αφορά την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ο κύριος Στάνοκ επισήμανε στην έκθεση το πιο βασικά στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εξέταση της ετοιμότητας του, Ευρωπα... Μαυροβουνίου για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, οικονομική διάρθρωση του Μαυροβουνίου. Πολύ σημαντικό θέμα. Την τελευταία διετία το Μαυροβούνιο ανέπτυξε τις τουριστικές υποδομές με αξιέπαινο τρόπο. Είναι πολύ καλές οι επιδόσεις του Μαυροβουνίου στον τομέα αυτό, αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι ο τουρισμός είναι ο μοναδικός σημαντικός κλάδος στη χώρα αυτή. Και άλλοι ε, κλάδοι είναι σημαντικοί που δυστυχώς τελευταία έχουν αποδυναμωθεί. Ήταν σημαντικοί τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά οικονομικοί κλάδοι τον τελευταίο καιρό έχουν ε, υποστεί μαρασμό. Βέβαια υπάρχουν και θετικά σημεία που θα μπορούσαμε να τονίσουμε και συμφωνώ με παρατήρηση του προλαλήσαντα ότι το κοινοβούλιο του Μοντενέγκρο χαρακτηρίζεται από μια ενότητα σε ό,τι αφορά σημαντικού στρατηγικού στόχου. Είναι ένα πολύ ζωηρό κοινοβούλιο. Για θέματα ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν συζητούσαμε όταν συζητούσαν το θέμα της προσχώρησης ε, στο ΝΑΤΟ ή σε άλλες διαδηλατικές ε, δομές. Το κοινοβούλιο του Μοντενέγκρου ήταν αρκετά συσπηρωμένο. Υπάρχει όμως πρόβλημα με τις μειονότητες. Παρόλο που οι μεγάλες μειονότητες προστατεύονται, αισθάνονται ασφαλείς και μπορούν να συμμετέχουν στην πολιτική και πολιτιστική ζωή. Προβλήματα υπάρχουν με τρεις κύριες μειονότητες, όπως φαίνεται και στις δύο εκθέσεις, και στην τελευταία του κυρίου Τάνοκ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόβλημα αντιμετωπίζουν τρεις μειονότητες, οι μειονότητες Ρωμά, Σκάλι και Αιγυπτιακή. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις παραδόσεις, γιατί δυστυχώς παραδοσιακά υπάρχει μια αναισθησία σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στο δημόσιο βίο. Αυτό είναι θέμα νοοτροπίας και καλό θα ήταν το Μαυροβούνιο να υιοθετήσει μια πιο ανεκτική νοοτροπία και φυσικά να δείξει μεγαλύτερη ανοχή και ως προς τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων. Συμφωνώ ότι το Μαυροβούνιο είναι μια χώρα που συμβάλλει στην σταθερότητα της, περι... περιοχής, έχει καλές σχέσεις γειτονίας με τις όμορες χώρες και θα πρότεινα Στη διαδικασία αυτή, στην προεταξιακή διαδικασία και στην πορεία προσχώρηση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιλύσει πρώτα το Μαυροβούνιο τα διασυνοριακά διαμεθοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει με την Κροατία. Αυτό όμως αφορά και την Κροατία. Η ε, κυρία Κοπά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω κι εγώ να συγχαρώ τον συνάδελφο Τάνοκ στην έκθεσή του και αυτό γιατί σε μια κρίσιμη στιγμή για όλη την πορεία της διεύρυνσης έχει σημασία τόσο η Επιτροπή όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στέλνει θετικά μηνύματα. Γι' αυτό η θέση πως οι διαπραγματεύσεις πρέπει να ξεκινήσουν το, το γρηγορότερο δυνατό είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η χώρα, το Μοντενέγκρο, έχει προχωρήσει πολύ τα τελευταία χρόνια. Προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν και δεν θα διαφωνήσω με τον συνάδελφο Ντανζάν ότι η επισήμανση για θέματα οργανωμένου εγκλήματος ή διαφθορά είναι σημαντικές και είναι αληθινές όμως για όλες σχεδόν τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Παρόλα αυτά η έκθεση με ισορροπημένο τρόπο εντοπίζει τα προβλήματα καθώς επίσης και για τα θέματα ελευθερίας γνώμης ή για την παράγραφο στην οποία αναφέρεται στις γυναίκες. Εδώ ίσως θα ήθελα μία εντονότερη διατύπωση για τα αυξημένα θύματα ενδοοικογενειακής βίας ε, στο Μαυροβούνιο καθώς και στην ανάγκη να υπάρξει μια εκστρατεία για τα δικαιώματα των γυναικών, ένα θέμα στο οποίο η χώρα ξεκινάει πραγματικά ε, αρκετά αργά. Ε, μία διαφωνία έχω να διατυπώσω για το θέμα του περιβάλλοντος. Ε, είναι αλήθεια ότι η χώρα έχει ένα τεράστιο δυναμικό ενεργειακό. Ε, έτσι όπως αναφέρονται όμως τα υδροηλεκτρικά έργα, ίσως να δημιουργούσαν πρόβλημα στο περιβάλλον και νομίζω ότι θα άξιζε μία αναφορά στις μεγάλες δυνατότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που έχει η χώρα. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρώ επίσης και την αναφορά του ε, στην, προτροπή του να λυθεί η συνοριακή διαφορά με την Κροατία με, με προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Γενικά είναι μια έκθεση που αντικατοπτρίζει πολύ καλά την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέναντι στο Μαυροβούνιο και θέλω για μία ακόμα φορά να τον συγχαρώ. Merci. Monsieur Τάλερ. Ευχαριστώ κύριο Στάλερ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον συνάδελφο Τάνοκ, τον εισηγητή μας, γιατί πιστεύω ότι η έκθεσή του είναι πραγματικά αξιόλογη και θα ήθελα να συμβάλλει σε ταχύτερη ενσωμάτωση του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Μαυροβούνιο ή είναι πολύ τυχερό, είναι πολύ έξυπνο, γιατί είναι η μόνη χώρα της περιοχής που δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα που να τον εμποδίζουν, να αυτή τη χώρα στο δρόμο της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο προβλήματα έχει, το Κωσυφοπαίδιο και το Μλάντι. Η Σερβία έχει μόνο δύο προβλήματα, το Μλάντιτς και το Κωσυφοπαίδιο. Η Βοσνία έχει πρόβλημα με την εσωτερική λειτουργία. Η Μακεδονία έχει πρόβλημα με την Ελλάδα. Το Κωσυφοπέδιο έχει επίση προβλήματα. Το Μαυροβούνιο είναι η μόνη χώρα που δεν έχει προβλήματα. Και άρα θα πρέπει να βοηθήσουμε αυτή τη χώρα να δράξει την ευκαιρία αυτή και να επιταχύνει την ε, πορεία ένταξη προ την Ευρωπαϊκή ένταξη, ε, Ένωση. Φυσικά αυτό συνδέεται και με την πολιτική βούληση αυτή τη χώρα, γιατί αν μια πολιτική δύναμη είναι παρούσα μια χώρα για πολύ καιρό στον ίδιο στο ίδιο πολιτικό περιβάλλον, ίσως δημιουργηθεί ένα, δημιουργηθεί ένα είδος αδράνειας και μια χαλάρωση της πολιτικής βουλής. Και αυτό είναι το πρόβλημα του, Μα, του Μαυροβουνίου, ότι δεν υπάρχει αρκετός πλουραλισμός. Δεν υπάρχει αρκετή ανοχή προς τις α, αντίθετες απόψεις, προς τις διαφορετικές απόψεις. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τις μειονότητες, αλλά αυτό οφείλεται και στην οτροπία που έχουν απέναντι στην κοινωνία των πολιτών. Γιατί πολύ συχνά η κοινωνία των πολιτών αντιμετωπίζεται ως ε, δημόσιος εχθρός. Κάτι που είναι ανόητο κατά τη γνώμη μου. Και ένα μεγάλο μέρος της βίας ε, στο Μαυροβούνιο οφείλεται στην καταστολή και στην καταπίεση, στον εκφοβισμό αυτών που καταγγέλουν περιπτώσεις δωροδοκίας ή οργανωμένου εγκλήματος. Όποιος καταγγέλει ε, ένα, μια περίπτωση διαφθοράς ή οργανωμένου εγκλήματος μπορεί να ξυλοκοπηθεί το ίδιο βράδυ που έκανε τις δηλώσεις. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε το Μαυροβούνιο να ανακτήσει την πολιτική βούληση και να επισπεύσει αυτή τη διαδικασία. Το Μαυροβούνιο αναφέρεται ως οικολογικό κράτος. Πολύ καλή πρόταση βέβαια αυτή, αλλά όποιος κάνει ένα ταξίδι στο Μαυροβούνιο διαπιστώνει ότι αυτά είναι μάλλον αγαθές προθέσεις. Στην πράξη δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Το Μαυροβούνιο θα πρέπει να έχει μια άγρια ομορφιά, αλλά ας επικεντρωθούμε περισσότερο στην ομορφιά παρά στο άγριο τμήμα αυτής. Ευχαριστώ. Merci, Monsieur Peterle. Ευχαριστώ κύριο Πέτερλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον συνάδελφο ε, Τάνοκ για την πολύ καλή και ρεαλιστική του έκθεση που είναι και αρκετά αισιόδοξη. Θα ήθελα όμως να συγχαρώ και το Μαυροβούνιο το ίδιο γιατί κατάφερε να προωθήσει μεταρρυθμίσεις που οδήγησαν στην ε, πολύ θετική αξιολόγησή του από τον εισηγητή μας τον κύριο Τάνοκ. Το Μαυροβούνιο πλησιάζει όλο και περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω ότι θα ενταχθεί σε αυτή το συντομότερο δυνατό με κάλυψαν οι προλαλήσαντες. Θα ήθελα απλώς να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με την ενταξιακή πορεία του Μαυροβουνίου και χαίρομαι που δεν υπάρχει καμία εσωτερική αντιπαράθεση ως προς την ανάγκη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτή η συσπήρωση και αυτή η ενότητα του Ευρωβουνίου υπέρ της ευρωπαϊκής προσχώρησης είναι πολύ σημαντικό. Δεν πρόκειται να σας καθυστερήσω άλλο γιατί οι συνάδελφοι με κάλυψαν και εγώ εκτιμώ ιδιαίτερο την πρόοδο που κάνουν οι χώρες στην ενταξιακή τους πορεία, όλες οι χώρες των Δυτικών Βαλκονίων, αλλά η πρόοδος του Μαυροβουνίου πιστεύω ότι θα επηρεάσει θετικά και τις άλλες χώρες της περιοχής. Merci. Pour la Commission européenne, Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω και εγώ το κείμενο του κυρίου Τάνε. Τάνοκ είναι βέβαια ένα έγγραφο του Κοινοβουλίου, δεν πρέπει να το σχολιάσουμε. Αλλά βλέπουμε ότι σε μεγάλο ποσοστό ευθυγραμμίζεται με την άποψη της Κομισιόν και τις σχετικές συστάσεις. Ακολουθούμε λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη ε, συζήτηση και περιμένουμε να δούμε την τελική διατύπωση του κειμένου. Ευχαριστώ κύριε Κούκαν. Με συγχωρείτε, έπρεπε να σας έχω δώσει το λόγο. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. nič ani ani čo by ευχαριστώ, πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι οι συνάδελφοί Έδωσα μια καλή εικόνα του Μαυροβουνίου στην Ευρώπη. Υπάρχουν δυνατότητες βέβαια για βελτίωση σε πολλούς τομείς, όπως παραδείγματος χάρη αφορά τα ΜΜΕ, έλλειψη ανοχής και ανεκτικότητας για ανεπίσημες απόψεις, διαφθορά ε, κλπ. Ταυτόχρονα θεωρώ ότι σήμερα μπορούμε να θεωρήσουμε το Μαυροβούλι μια χώρα η οποία βάσει αυτής της έκθεσης έχει πάρει την, ε, το καθεστώς της υποψήφιας χώρας και περιμένουμε ποια θα είναι η ημερομηνία έναρξης των διαπραγματεύσεων. Ελπίζω να μην χρειαστεί να περιμένει τόσο πολύ όσο άλλες υποψήφιες χώρες και θα πρέπει νομίζω να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας στο Μαυροβούνιο ούτω ώστε τα θέματα που παραμένουν εκκρεμή να επιληθούν το γλυγορότερο δυνατόν Ούτως ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν πραγματικά οι διαπραγματεύσει. Μέσα σε αυτό το πνεύμα είναι ρεαλιστικό το κείμενο του κυρίου Τάνο και θα ήθελα να σας πω ότι πραγματικά σε σχέση με τις άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων το Μαυροβίνο έχει τις τα λιγότερα προβλήματα και ο συνόλογος Τάν ε, αναρωτήθηκε κατά πόσον αυτό είναι εξυπνάδα μέρος τους ή τύχη. Και τα δύο λίγο θα έλεγα. Γιατί πραγματικά εκμεταλλεύονται όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν προς όφελός τους και μπορώ γι' αυτό να συμφωνήσω με το έγγραφο όπως έχει υποβληθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Στάνοκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όταν η ομάδα μου αγόρασε εντό εισαγωγικών την έκθεση του Μαυροβουνίου, ε, είχα πραγματικά την εντύπωση ότι θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα από ότι για κάποιου άλλου ε, γείτονε. Και μπορώ να συμφωνήσω με τον κύριο Κούκαν που είναι και εμπειρογνώμονα του θέματο και ο κύριο Στάλλα, επίση ε, διακεκριμένο μέλο τη ε, Υπουργό Εξωτερικών είναι σωστό ότι το Μαυροβούνιο είναι η λιγότερο πληματική χώρα τη περιοχή και θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Και εγώ είμαι μεταξύ αυτών που είναι υπέρ τη ε, αρχή τη κοπηλοδρομία. ότι θα πρέπει δηλαδή όσον αφορά τη διαδικασία ένταξης να προχωρήσουν αμέσως μετά την Κροατία που θα είναι η πρώτη. Και <clears throat> ανοιχτή όλα τα σχόλια που έκαναν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ τον κύριο Ντονζό, τον κύριο Βάιγκαλ, την κυρία Καπά που τόνισε το θέμα των δικαιωμάτων των γυναικών που δεν γνωρίζω τι λεπτομέρειες μου και αν έχει πραγματικά κάποια σχόλια για το θέμα αυτό θα ήμουν πολύ ευγνώμη να μου τα υποβάλει. Επίσης, ο περάσινος συνάδελφος που αναφέρθηκε στο θέμα του σεξουαλικού προσανατολισμού και τα δικαιώματα των αφιλοφίλων. Δεν συμφωνώ όμως ότι ελέγχθη για την ε, υπηκότητα, γιατί κάθε ε, κυρίαρχο κράτος ε, πρέπει να έχει το δικαίωμα να δίνει την υπηκότητά του όπου θέλει. Και στη χώρα μου. Αν ε, έχει κανένα χρήματα μπορώ να αγοράσει ε, τη δυνατότητα να εγκατασταθεί εκεί. Το μόνο πρόβλημα είναι το θέμα της ελεύθερης κυκλοφορίας ε, όταν είναι κάποιος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή άμα δίνουν ε, χιλιάδες διαβατήρια σε ανθρώπους που έρχονται από τέτοιες χώρες, αυτό θα είναι προβληματικό όσον αφορά την κινητικότητά τους προς άλλα κράτη-μέλη. Και θα πρέπει βέβαια τότε να σχολιάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν είναι θέμα μετανάστευσης. Ε, όσον δεν φτάσει εκεί όμως, το μαυροβούνιο είναι και αυτό κυρίαρχο και μπορεί να δώσει την υποκότητά του όπου θέλει. Εκτό αν κάποιο πει ότι αυτοί είναι καταζητούμενοι εγκληματίε. Όχι. το όψεις και περιπτώσει να ακούσαμε ποτέ δεν ήταν το μακροβούνο ενάντια στο θέμα της ε, έκδοσης κάποιων ε, πολιτών. Από ξέρω, ο, πρόσφατα υπέγραψε το Παυροβούνιο μια διμερή συμφωνία έκδοση με τη Σερβία. γιατί ελέγχθη ότι κάποιοι από τον τομέα του οργανωμένου εγκλήματος είχαν καταφύγει στο Μαυροβούνιο λόγω της υπηκότητας που είχαν πάρει. Από τώρα ξέρω ότι αυτή η νέα συμφωνία έκδοση δεν έχει ακόμα επικυρωθεί και από τα δύο κοινοβούλια, αλλά υπάρχει τέλο πάντων. Και υπάρχει και μία που ισχύει με την Κροατία, που ισχύει και για τους ίδιους πολίτες. Όπου υπάρχει δηλαδή αυτή η διμερή συμφωνία, δεν ισχύει αυτό το θέμα. Και το θέμα του περιβάλλοντος που έθιξαν διάφοροι συνάδελφοι. Ε, ξέρουμε διάφορους που μπορούν να βελτιώσουν ε, ποιότητα του νερού, ποιότητα του αέρα και αν έχετε συγκεκριμένα στοιχεία σας παρακαλώ να μου τα υποβάλλετε σε λεπτομέρειες. Κατά τα άλλα, ε, ήμουν πολύ ικανοποιημένο για τον τρόπο με τον οποίο έγινε δεκτή η έκθεσή μου από την Επιτροπή και οπωσδήποτε δεν είναι πιο αντιλεγόμενη από εκείνες που έχουμε μπροστά μας στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών λίγη στις 14 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης, Μαύρη Θάλασσα. Συζήτηση για τις τροπολογίες. Πάνω συνέξη πρωτοβουλίας για στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Μαύρη Θάλασσα. Ο εισηγητής είναι ο κύριος Ουγγουρεάνο. Είχαμε στις 9 Νοεμβρίου μια πρώτη συζήτηση του θέματος. 131 τροπολογίες υπευλήθησαν η Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου και Βιομηχανία και η Επιτροπή Έρευνα και ενέργεια ήδη υπέβαλαν τι γνωμοδοτήσει του και η γνωμοδότηση τη επιτροπή περιφερειακή Ανάπτυξη θα υιοθετηθεί σήμερα. Το λόγο για τον κύριο Σουμπουριανού για να σχολιάσει τι διάφορε τροπολογίε του σχέδιου αυτό ψηφίσματο. Ευχαριστώ πρόεδρε Πράγματι υπευλήθησαν 131 τροπολογίες. Και με ικανοποίηση είδα ότι σχεδόν όλες είναι επικοδομητικές. Υπάρχει μια γενική συνένεση όσον αφορά την γενική προσέγγιση, ότι χρειάζεται δηλαδή περισσότερη παρακολουθήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μια πολιτική σαν μια σωστή κοινωνική πολιτική. Υπάρχει και συνένεση μεταξύ των ε, πολιτικών ομάδων για τις γενικές ε, τροπολογίες, οι περισσότερες τροπολογίες από το ΕΛΚ, τους σοσιαλιστές, ε, τους φιλελεύθερους και ακόμη μάλιστα και από τους πράσινους ορισμένοι είναι επικοδομικές και αποδεκτές. Υπάρχουν και άλλα θέματα πάνω στα οποία προτείνουν κάποιους συμβιβασμούς για να υπάρχει μια πιο καλή οργάνωση του κειμένου, να αποφευχθούν οι αντιφάσεις και οι επαναλήψεις. Τι πιο στο τομείς συμβασμών είναι η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατάσταση του περιβάλλοντος και θέματα ενέργειας και υποδομές. Αύριο λαμβάνει χώρα μία συνάντηση με τους κοιόδης ηγητές στις 12.30 αν δεν κάνω λάθος και ελπίζω θα μπορέσουμε εκεί να συζητήσουμε τις τροπολογίες και τις συμβαστικές τροπολογίες για να βρούμε ένα κοινό έδαφος. Βέβαια, υπάρχουν και μερικές ε, τροπολογίες που δεν μπορώ να δεχτώ. Καταρχήν, την τροπολογία που προτείνει την θεσμοποίηση ή την δημιουργία νέων δομών στην περιοχή του Ξινού Πόντου, είναι η την δημιουργια νεων δομων στην περιοχη του φξινου ποντου ειναι η τροπολογια 29, για τη δημιουργία μιας ένωσης, η 56, για μια τριμερή ε, δομή μεταξύ Τουρκίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας επίσης. Δεν χρειάζονται νέες δομές, δεν χρειάζονται νέα θεσμικά όργανα στην περιοχή του ευθύνου Πόντου υπάρχουν ήδη πάρα πολλε οργανώσεις εκεί. Υπάρχουν πάρα πολλε πρωτοβουλιε Εγώ θεωρώ ότι η δημιουργία νέων ε, δομών θα είναι εις βάρος ε, της εφαρμογής αυτών που έχουμε όσον αφορά την τριμερή σχέση Τουρκίας δηλαδή και Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ τόνισα ήδη τη σημασία της Ρωσίας και της Τουρκίας στην περιοχή. Αλλά είναι δύσκολο να δεχθούμε μια τροπολογία που κατά κάποιο τρόπο αποκλεί άλλους ενδιαφερόμενους από την περιοχή εκεί για μια περιφερειακή συνεργασία. Και η δεύτερη ομάδα είναι οι τροπολογίες 38 και 39 που προτείνουν τη διαγραφή ορισμένων διατάξεων για μια ξεχωριστή γραμμή του προπολογισμού για την πολιτική στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, του Ευξηνοπόντου. Αυτό είναι ένα κεντρικό θέμα της έκθεσής μου, να υπάρχει δηλαδή αυτή η ξεχωριστή γραμμή στο προπολογισμό. Με ενέπνευσαν εδώ και οι συνάδελφοι που εργάστηκαν για την στρατηγική για την Βαλτική που προβλέπεται και εκεί επίσης μια ξεχωριστή γραμμή στο προπολογισμό και θα ήθελα να σας προτείνω επίσης ότι η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωση στον Ευξοπόντο είναι καταγραμματισμένη και γι' αυτό χρειάζεται κάτι να γίνει. Επίσης θεωρώ ότι είναι δύσκολο να δεχτώ κάποιε τροπολογίε που υπέβαλε η FTN και η TCR που έχουν σαν στόχο τον περιορισμό του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή του αυξήνου πόντου. Με ενδιαφέρον θα ακούσω τα σχόλιά σας και όπως σας είπα θα συνεργαστώ αύριο με τους σκιώδεις και τονίζοντας, θα ήθελα, ε, το συγγνώμη, θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά την γενική γραμμή που πήρε η πλειοψηφία και να σα ευχαριστήσω για τα σχόλιά σας. Merci, σας ευχαριστώ κύριε Σιγητό και Καζάκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή το να αναζωογονήσουμε την ε, Μαύρη Θάλασσα με τέτοια μέτρα μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο συζητητής γνωμοδότησης στα πλαίσια της Επιτροπής Σύντα για την Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Εύξηνο θα ήθελα να τονίσω κάποια συγκεκριμένα κύρια θέματα που θα ήθελα να συμμεριστώ μαζί σας. Καταρχήν, όπως σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή, πλήγει και η περιοχή της ε, Μαύρης από την οικονομική κρίση, η οποία μείωσε το ποσοστό ανάπτυξη που υπήρχε τη τάξη του 6% και πιστεύουμε ότι εάν ε, δυναμωθούν τώρα οι τραπεζικοί και δημοσιονομικοί κανόνες, θα μπορέσει να ξανααρχίσει να αναπτύσσεται η συνεργασία σε Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητη. Υπάρχουν όμως διάφορες ε, περιφερειακές ε, διμερείς ε, συμφωνίες συνεργασίας και αυτό κινδυνεύει να κατακαιρματίσει τις προσπάθειες και να υπάρχουν επικαλύψεις διαφόρων χρηματοδοτήσεων. Η στρατηγική του ξένου πόντου θα πρέπει να οικοδομηθεί πάνω στις κεκτημένες εμπειρίες από άλλες περιοχές, την Βαλτική, τα Βαλκάνια, τον, του Δούναβη, χωρίς να τονίσουμε κάποια περιοχή περισσότερο από την άλλη. Η συνεργασία με άλλες τοπικές οργανώσεις, όπως παραδείγματος η Οργάνωση για την Οικονομική Ανάπτυξη του Πόντου, είναι και αυτό σημαντικό. Να απτυχθούν προγράμματα υποδομής για την περιοχή. Είναι επίσης σημαντικό. Ιδίως έχω εδώ κατά νου το ενεργειακά προγράμματα από το Ναμπούκοφ, η ανάπτυξη των χερσαίων και θαλασσίων οδών που θα μπορούσαν να διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές στην περιοχή εκεί και επίσης να αυξηθεί το δυναμικό των ε, λιμένων Κωνστάτσα και Τζουμπάλα είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν και δύο χώρες που δεν είναι ακόμα μέρη της διεθνούς, ε, του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου στην περιοχή εκεί και εγώ θα επιθυμούσα όλες τις χώρες του ευξήνου πόντου να γίνουν μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης. Ο εισηγητής θέλησε να προσθέσει τις τροπολογίες που αφορούν τη συνεργασία με άλλους ε, φορείς, ε, Παραδείγματο όσον αφορά τους ε, λιμένες της Κωνσταντσα και της Βάρνα, και όσον αφορά την, το Δούναβι, συμφωνώ με τον κύριο Πάσκου. Πιστεύω ότι η περιοχή του Δούναβι τονίζει την γεωστρατηγική σημασία του αυξήνου πόντου και ότι υπάρχει και ένα ειδικό γεωγραφικό ενδιαφέρον. Τέλος, υποστηρίζω την άποψη των κ. Βάγκελ και που ζητούν να διευκολυνθεί το καθεστώς θεωρήσεων διαβατηρίου έναντι των χρόνων της περιοχής. Ελπίζω ότι η στρατηγική αυτή θα καλύψει καλύτερα τις προσδοκίες μας για την περιοχή του Ευξήνου Πόντου και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Κόπα. Ε, θέλω να πω μερικά σημεία για την περιοχή του Εύξηνου Πόντου, μια ξεχωριστή γεωγραφική περιοχή, πλούσια σε φυσικούς πόρους και εξαιρετική γεωγραφική θέση. Είναι μια περιοχή όμως που υπάρχουν ανεπίλητες παγωμένες διενέξεις, αλλά και πολλά άλλα θέματα όπως οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η παράνομη μετανάστευση, το οργανωμένο έγκλημα και άλλα. Η έκθεση του εισηγητή του κύριου ε, Ουγγουρεάνου προσπαθεί να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις πτυχές ε, με μεγάλη επιτυχία και θέλω να τον συγχαρώ για το κείμενο που μας κατέθεσε. Η περιοχή είναι μια περιοχή με μεγάλο ενεργειακό δυναμικό και για μας είναι πολύ σημαντική η ενίσχυση της ενεργειακής σταθερότητας. Στην έκθεσή του, ο τονίζει τα πλονεκτήματα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συνεργασία της σε αυτή την περιοχή, καθώς και το ρόλο της Ένωσης ε, στο, ε, στην συνεργασία στον ενεργειακό τομέα και στη δημιουργία μιας ζώνης ελευθέρων συναλλαγών. Αυτό που νομίζουμε είναι ότι χρειάζεται να ενισχυθεί η έκθεση στα ζητήματα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτή ήταν η κατεύθυνση των δικών μου τροπολογιών καθώς επίσης και να τονιστεί ότι η συνεργασία με την Ένωση θα συνεισφέρει στη βελτίωση της κατάστασης στις χώρες αυτές, είτε οικονομικά είτε πολιτικά, με την ενίσχυση της δημοκρατίας, την καταπολέμηση της διαφθοράς κτλ. Αυτή ήταν η κατεύθυνση των τροπολογιών μου και πάλι να συγχαρώ τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Uh, uh, Ο κ. Σεβερά, σας ευχαριστώ πρόεδρε. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην προσέγγιση της ε, περιοχής, κάποια προκατάληψη η οποία λέει ότι θα μπορούσε κάποιο να αναπτύξει την οικονομική συνεργασία, την περιβε... περιβαλλοντική συνεργασία και άλλες συνεργασίες χωρίς να ασχοληθεί με τα θέματα της ασφάλειας. Πρόσφατα είχα επισκεφτεί την περιοχή και αναγνώρισα ότι πράγματι εφόσον τα θέματα της ασφάλειας δεν αντιμετωπιστούν σωστά, δεν μπορούμε να προβλέψουμε την εξέλιξη των άλλων διαστάσεων συνεργασίας στην περιοχή. Γι' αυτό πιστεύω και μάλιστα να προσθέσω ότι αν πρόκειται για θέματα ασφαλείας, ξαφνικά οι δύο από τις χώρες περιοχής διστάζουν πάρα πολύ να έρθουν σε επαφή μαζί μας. Και ακριβώ αυτέ οι δύο χώρε είναι η Ρωσία και η Τουρκία. Βρίσκουμε, βρισκόμαστε λοιπόν σε κάποιο φαύλο κύκλο. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο εισηγητή να ξαναμελετήσει την άποψή του όσον αφορά μία από τις τροπολογίες που αφορά την ανάγκη δρέωσης της ε, μορφής συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ρωσίας και Τουρκίας όχι να αποκλειστούν οι άλλοι, αλλά ακριβώς για να μπορούμε να δημιουργήσουμε το, το σωστό περιβάλλον για να συμπεριληφθούν και οι άλλοι. Γιατί αν θέλουμε να είμαστε πολιτικά σωστά και πούμε ότι εμείς δεν κάνουμε διακρίσεις μεταξύ των εταίρων μας, δεν θα είμαστε όσο αποτελεσματικοί θα έπρεπε. Αυτή είναι η σημασία λοιπόν μια από τις τροπολογίες μου. Και θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι ακριβώς πρόσφατα στο επίπεδο της δικής μου πολιτικής ομάδας Είχαμε μια τέτοια διάσκεψη και υπάρχουν πολλές πιθανότητες αυτού του τύπου η προσέγγιση να είναι επικοδομητική. Όχι για να αποκλείσουμε κάποιον, επαναλαμβάνω, αλλά για να μπορέσουμε ακριβώ να καταστήσουμε τελικά να συμπεριλάβουμε τους πάντες. Γιατί αυτοί οι δύο εταίροι που αυτοαποκλείονται για διάφορους λόγους θα πρέπει εμείς να φροντίσουμε να τους εντάξουμε πριν έχουμε μια πιο ευρία διάσκεψη. Και η τελευταία μου παρατήρηση είναι ακριβώς σε σχέση με μια δεύτερη, τη δεύτερη τροπολογία στην οποία αναφέρθηκε ο εισηγητής, ο κ. Σουγκουριάνο, ακριβώς αυτή η ιδέα της ε, ένωσης εξήνου πόντου. Ίσως κάτι θα μπορούσαμε να αλλάξουμε όσον αφορά αυτή την ονομασία αν θέλετε. Αλλά παρόλο που συμφωνώ με την εισηγητή ότι υπάρχουν ήδη πάρα πολλέ πρωτοβουλίε, πάρα πολλέ οργανώσει και δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτα, από την άλλη μεριά δεν υπάρχει καμία τέτοια οργάνωση στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει το ρόλο πρωταγωνιστή. Εάν λοιπόν δούμε κάτι όπως εκείνο για τη σχέση με την Μεσόγειο, μια ένωση για τη Μεσόγειο, μπορούμε κάτι παρόμοιο να έχουμε για τον εύξηνο πόντο, για να έχουμε έτσι μια πολιτική υπερδομή αν θέλετε μόνο και μόνο για να ενδυναμώσουμε τη στρατηγική μας που χρειάζεται και που θα αντικαταστήσει νομίζω τη σημερινή συνεργία που είναι αυτή καθ' αυτή η αναγνώριση ότι λείπει η στρατηγική. Κύριος Κυριλόφ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Γκουρεάνου για μια πληρέστατη έκθεση και για τις προσπάθειες που έκανε η έκθεση αυτή να είναι αντικειμενική. Έχω κάποια σχόλια σε αυτά τα οποία άκουσα προηγουμένως. Θα ήθελα να πω ότι η προσπάθεια είναι δύσκολη στενότερη συνεργασία στην περιοχή είναι κάτι το πολύ δύσκολο. Ξέρετε ότι υπήρχαν τέσσερις χώρες κάποτε, τώρα είναι σχεδόν οχτώ. Μία από τις χώρες αυτές θα έλεγε ότι είναι και πάνω από οχτώ. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Κάποιες από τις χώρες δεν είναι πάρα πολύ ευχαριστημένες από τις πολιτικές τις οποίες επιδιώκουμε. Για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις πολιτικές αυτές, θα πρέπει να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον τους και να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε μία από αυτές. Η Μαύρη Θάλασσα είναι μια σκληρή θάλασσα θα έλεγα, επικίνδυνη. Έχουμε πολύ σοβαρά ατυχήματα. Χτες υπήρξε μια σύγκρουση πλοίων, βυθίστηκε ένα πλοίο, πνίγηκαν έξι ναυτικοί, τέσσερις σώθηκαν με τη βοήθεια των βουλγαρικών αρχών. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια ειδική παράγραφο στην έκθεση αυτή για τέτοιου είδους θέματα, γιατί αυτά τα θέματα αφορούν όλες τις χώρες και εγώ έχω καταθέσει μία τροπολογία επιμένοντας τη σημασία που έχει η διάσωση στη θάλασσα. Έκκλησή μου είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε λοιπόν πράγματα, θέματα τα οποία σε ένα πρώτο επίπεδο θα πείσουν όλες τις χώρες να συνεισφέρουν με την δραστήρια βέβαια στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Σούς. Πρόεδρε, Ήδη μία φορά συζητήσαμε αναλυτικά την στρατηγική της Μαύρης Θάλασσας και είδαμε να υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία. Γι' αυτό εγώ θα θέλω να αναφερθώ στις τροπολογίες και στις ε, ε, διευκρινήσεις και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Κουριάνο, ότι θεώρησε τις τροπολογίες μας ε, επικοδομικές και είπε ότι σε μεγάλο ποσοστό θα τις συμπεριλάβει στην έκθεσή του. Εμείς θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της χρηματοδότησης μικρών αναπτυσσιακών προγραμμάτων. Τα λεγόμενα people to people. Από τους ανθρώπους και τους ανθρώπους. Δηλαδή ενδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενίσχυση μη κυβερνητικών οργανώσεων, καταλληλών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Θα πρέπει όλοι αυτοί να συμπεριληφθούν στην εφαρμογή της αρχικής του ευξήνου πόντου Και απ' την άλλη θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις διαμάχες που εξακολουθούν να υπάρχουν, να τις εντάξουμε σε ένα πρόγραμμα έγκυρης προειδοποίησης για να μπορούσαμε να τις επιλύουμε έγκαιρα και να μην υπάρχει <clears throat> όξυνση. Επίσης, όσον αφορά το θέμα της ε, ενεργειακής πολιτικής, Ναμπούκο, South Stream, και επίσης θα πρέπει να φροντίσουμε να ε, σταθεροποιήσουμε υπάρχοντα δίκτυα στον ε, πανεπιστημιακό τομέα, στον φοιτητικό τομέα και να υπάρχει και ένα Ινστιτούτο για ευρωπαϊκές ε, μελέτες που χρειαζόμαστε στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Αν όλα αυτά συμπεριληφθούν, τότε η έκθεση αυτή θα έχει το σωστό Ε, Ευχαριστώ. Σεβιτς. Λέω κύριο Σίβιετς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η πρωτοβουλία για τη συζήτηση αυτή είναι πάρα πολύ θετική. Βέβαια δεν συζητάμε για πρώτη φορά το θέμα της στρατηγικής για τη Μαύρη Θάλασσα υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε γιατί είναι περίπλοκη η περιοχή. Όταν προσπαθούμε να φέρουμε κοντά κάποιες χώρες από την περιοχή είναι σαν να φέρνουμε σε επαφή το νερό και τη φωτιά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να λύσει τα προβλήματα της περιοχής στην κατάσταση που βρίσκεται δεν μπορεί. Υπάρχει κι άλλο ένα στοιχείο που δεν έχει αναφερθεί στην έκθεση αλλά έχει μεγάλη σημασία και αφορά τη δημιουργία δικτύων ανάμεσα στις χώρες της περιοχής. Διακοινοβουλευτική συνεργασία σαν παράδειγμα. Υπάρχει ένας θεσμός που ονομάζεται Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Μαύρης Θάλασσας. Είναι μια οργάνωση η οποία έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία θα τα ονόμαζα, πώς να το πω, είναι λίγο ιδιόμορφη. Εκφράζει θα έλεγα κάποιες αντιλήψεις οι οποίες ανήκουν στο παρελθόν όταν η Σοβιετική Ένωση κυριαρχούσε στην περιοχή. Η οργάνωση αυτή ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακόμη και με αποστολή ad hoc αντιπροσωπείας Και έλαβα το λόγο αυτό το θέμα γιατί στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία ως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχα... ήμουν αρμόδιος για τις επαφές με αυτή την οργάνωση. Και δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη, αλλά θα ήθελα να σημειώσω, να επισημάνω ότι έχουμε φοβερές καθυστερήσεις ε, στην πολιτική αυτή, αν δεν ενισχύουμε τις κοινοβουλευτικές επαφές. Και μερικέ φορέ έχουμε κάποιες φήμες που δεν ανταποκρί... ακούμε κάποιε φήμε που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στο τίτλο του εγγράφου αυτού λέγονται τα πάντα. Αναφερόμαστε στη στρατηγική της Μαύρης Θάλασσας Πρόκειται για μια περιοχή όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση επιγόντως χρειάζεται μια στρατηγική σε βάθος. Αυτό είναι ο μόνος δρόμος αν θέλετε έτσι ώστε η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας να γίνει ένα τμήμα της Ευρώπης, ένα τμήμα τουλάχιστον του κόσμου όπου η Ένωση να παίζει σημαντικό ρόλο ένα ρόλο ο οποίος θα βοηθάει και την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την περιοχή κυρίως. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Ίσως τελικά οι δυνατότητες που έχουμε στην περιοχή είναι περισσότερες ε, από τις άλλες περιοχές. Έχουμε τρεις χώρες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούν να βοηθήσουν έτσι ώστε να πετύχουμε τους κοινούς μας στόχους να πείσουμε δηλαδή για μια βαθύτερη ενσωμάτωση της περιοχής αυτής στην ευρύτερη περιοχή κοινών αξιών σεβασμού ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών. Νομίζω ότι κάτι το οποίο υπογραμμίζεται σωστά στην έκθεση του κυρίου Γκουρεάνου είναι ότι η περιοχή αυτή δεν είναι απλά μια οικονομική περιοχή, δεν είναι ένα οικονομικό πρόγραμμα το οποίο θα προωθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μας ενδιαφέρει η περιοχή αυτή γιατί έχουμε οικονομικά ή άλλα συμφέροντα. Αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε είναι να συμμεριστούμε με τις χώρες της περιοχής τις αξίες τις οποίες πρεσβεύουμε. Συνεπώς, οι χώρες της περιοχής και οι λαοί της περιοχής θα πρέπει να συνεισφέρουν στην ε, επίλυση των διεθνών διαφορών και των προβλημάτων που υπάρχουν, ιδιαίτερα των προβλημάτων αυτών που δεν μπορούν να ξεπεραστούν εάν δεν υπάρξει συμμετοχή των λεγόμενων περιφερειακών χωρών. Να υπογραμμίσω και άλλο ένα θέμα το οποίο τίθεται ίσως όχι πρόβλημα, αλλά κάτι το οποίο χαρακτηρίζει μια κάποια έλλειψη. Ο διαπολιτισμικός διαθρησκευτικός διάλογος είναι απόν και πρέπει να προωθηθεί. Ο διάλογος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πρότυπο συνεργασίας και με άλλες χώρες. Συμφωνώ με τον κύριο Κάζακ, ο οποίος είπε ότι η απελευθέρωση του καθεστώτος χορήγησης θεωρήσεων είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να προωθήσει τις δημοκρατικές διαδικασίες στην περιοχή. Το καθεστώς απελευθέρωσης των θεωρήσεων είναι σαφώς ότι θα φέρει τις χώρες πιο κοντά στις ευρωπαϊκές αξίες. Και τώρα μία τελευταία παρατήρηση να μου επιτρέψετε. Αυτή η περιφερειακή πρωτοβουλία θα πρέπει κυρίως να αντικατοπτρίζει τις δικές μας αξίες, τις αξίες του κράτους δικαίου, του σεβασμού της διεθνούς τάξης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ογκουρεάνου απαντά. Θα είμαι σύντομος. Υπάρχουν πολλά πάνω στα οποία μπορεί να σχολιάσει κανείς. Καταρχάς ευχαριστώ όλους για τις εξαιρετικές τους παρατηρήσεις που δείχνουν την ποιότητα της συζήτησης. Ξεκινώ με τις παρατηρήσεις του κυρίου Καζάκ Το έγγραφο της ΣΥΝΤΑ είναι κάτι το οποίο θα έλεγα παρουσιάζει πολλά θετικά και θα μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε ε, τις παρατηρήσεις που περιλαμβάνει η κυρία Καζάκ με πολύ σωστό τρόπο για τη χρησιμότητα του Ναμπούκο για το κοινοτικό πλαίσιο που πρέπει να μετατραπεί σε περιφερειακό πλαίσιο και οι παρατηρήσεις της κυρίας Κοπά για τα ανθρώπινα συμπεράσματα πρέπει να ληφθούν σοβαρά, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συγγνώμη, πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Σημειώνω επίσης αυτά που είπε και ο κύριος Σεβερίν. Έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση γύρω από τα θέματα αυτά. Όταν αναφέρεται κανείς για το τρίγωνο Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας-Ρωσίας, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί του ότι η Ρωσία και η Τουρκία είναι οι μεγάλες ε, δυνάμεις της περιοχής, αλλά ταυτόχρονα δύο και από τα μεγάλα προβλήματα της περιοχής. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή αντίληψη καταστεί στη Μαύρη Θάλασσα λειτουργική, τότε η Ρωσία και η Τουρκία θα παίξουν το ρόλο που τους αναλογεί. Ψυχολογικά τώρα, Διαρωτώ με αν και οι άλλες χώρες της περιοχής θεωρήσουν ότι περιθωριοποιούνται αυτή τη στιγμή η συνεργασία Τουρκίας, Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης πάρει μια συγκεκριμένη μορφή. Σχετικά με την Ένωση της Μαύρης Θάλασσας, συμφωνώ με τον κύριο Σεβερίνη, είναι μια άλλη συζήτηση. Δεν ξέρω αν η Ένωση για τη Μεσόγειο θα μπορούσε να ονομαστεί στη συγκεκριμένη φάση σαν success story, αλλά πάντως ε, δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Νομίζω ότι δεν μπορούμε εμείς να περάσουμε σε μια ένωση της Μαύρης Θάλασσας αν δεν οικοδομήσουμε τις βασικές αξίες γύρω από τον τρόπο με τον οποίο η Ένωση αντιμετωπίζει την περιοχή και έχει πάρα πολύ δίκιο ο, ο κύριος Σεβερίν. Αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι αρκετά. Να χαιρετήσω και τις παρατηρήσεις του κυρίου Κυριλόφ για την ασφάλεια στη θάλασσα. Οι τροπολογίες του είναι εξαιρετικές. Και να συμφωνήσω επίσης και με τον κύριο Σούλτς για την ε, βοήθεια για την ανάπτυξη. Αν δεν κάνω λάθος, άκουσα τον κύριο Σίβιετς να μιλάει για κοινοβουλευτική συνεργασία. Εφόσον αυτά τα οποία είπε ισχύουν, πρέπει να αναφερθούμε στην ομάδα αυτή των χωρών στην παράγραφο 7 της πρότασής μας. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Βάιγκελ για τις παρατηρήσεις του. Η αλήθεια είναι ότι η πραγματικότητα τώρα είναι ουσιαστικά μια έλλειψη, ένα κενό ουσιαστικής πολιτικής της Ένωσης απέναντι στην περιοχή. Δυστυχώς εκεί βρισκόμαστε τώρα. και θα δεχτώ την τροπολογία του για τη βελτίωση του καθεστώτος χορήγησης θεωρήσεων στους κατοίκους των χωρών της περιοχής. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Σας θυμίζω ότι η ψηφοφορία θα γίνει την 5η 9 Δεκεμβρίου και το επόμενο θέμα τώρα στην ημερήσια διάταξη αφορά τη Λιβύη. Η συγγήτρια είναι η κυρία Γκόμες, η οποία όμως θα έρθει όπου να είναι, σε πέντε λεπτά. Συνεπώς σας προτείνω να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Okay. compris.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 Συνεχίζουμε. Μόλις κατέθεσε και η κυρία Γκόμες. Χωρίς άλλη λοιπόν καθυστέρηση. Σας δίνω το λόγο κυρία Γκόμες. Merci, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας είμαι ευγνώμων για την υπομονή σας και την αναμονή. Το σχέδιο σύστασης που εκπώνησα και που θα συζητήσουμε και περιμένω με αδημονία τα σχόλια των σκιωδών εισηγητών των διαφόρων ομάδων έχει ως σκοπό να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται αυτή τη στιγμή μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ελληνικών Αρχών προς εκπλήρωση μιας εντολής που εμείς ακόμη δεν την έχουμε δει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρά τις επανειλημμένες μας εκκλήσεις και αιμονή να την εξετάσουμε. Φαντάζομαι θα ληφθεί απόφαση σύντομα, αλλά την εντολή αυτή δεν έχουμε δει. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι το περιεχόμενό της. Και παρά τη επαφές που είχαμε με τις αρχές της Λιβύης στήριξα το σχέδιο σύστασης στις πληροφορίες που συγκέντρωσα εγώ μετά από ταξίδι που πραγματοποίησα στη Λιβύη μαζί με την προσωπία του Μαγκρέμπ με επικεφαλή τον Αντώνιο Παντσέρη. Και Αντώνιο φαντάζομαι θα σας ενημερώσει εντός ολίγου για τις εντυπώσεις από την αποστολή αυτή. Είχαμε μία κάπως αμήχανη αφετηρία, αλλά έγιναν πολλές ενημερωτικές συναντήσεις και είχαμε αρκετά αφέλεις και αθώες. Εμείς είμαστε πολύ αφέλεις και αθώοι στις συζητήσεις. Πάντως, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παρατήσει τη Λιβύη. Έχουμε πολύ σημαντικές σχέσεις με τη χώρα αυτή και όχι μόνο κάποιες χώρες μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο έχει σχέσεις με την Λιβύη. Και το διακύβευμα αυτών των σχέσεων είναι τεράστιο. Αφορά την ενεργειακή μας ασφάλεια. Αφορά τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών την προστασία των προσφύγων και των ετούν τον άσυλο. Καλό θα λοιπόν να βοηθήσουμε, να ενθαρρύνουμε τη Λιβύη να εξελιχθεί πολιτικά και να γίνει σταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή. Και επίσης να συμβάλλει στην αναχέτηση των κλιματικών αλλαγών. Όπως είπα και στο σχέδιό μου, έχουμε να κάνουμε μια χώρα που είναι ιδιάζουσα. Είναι δικτατορικό το καθεστώς, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι ανέδοτο. Έχει συζητήσει μαζί μας, έχει συνάψει και συμφωνίες με κάποιες χώρες μέλη, τη Γαλλία και την Ιταλία κυρίως. Έχει στενές σχέσεις με χώρες όπως η Μάλτα. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να κάνουμε σαν να μην υπάρχει η Λιβύη. υπάρχει και είναι σημαντική και για την ασφάλειά μας και για τη διαχείριση πολλών ζητημάτων που μας απασχολούν. Θα πρέπει όμως να θέσουμε τους σωστούς όρους και να υποβάλουμε τα σωστά αιτήματα και να υποβάλουμε τις σωστές απαιτήσει και νομίζω ότι είναι πρόθυμη να μας ακούσει η Λιβύη. Ένα σημαντικό σημείο είναι ότι θα πρέπει καταρχήν να πείσουμε το Συμβούλιο να αποσύρει το αίτημα για τη συμφωνία επανεισδοχής με τη Λιβύη. Όχι επειδή δεν θα συμφωνήσουν ουδέποτε οι Λίβοι για τη συμφωνία αυτή, όπως και το Μαράκο και η Τουρκία, αλλά γιατί το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίφαση με τις δικές μας αρχές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πώς μπορούμε να ζητούμε επανειστοχή για μετανάστες από μια χώρα που χρησιμοποιεί εκτεταμένα τη θανατική ποινή, που δεν χαρακτηρίζεται από κράτος δικαίου, αλλά από κυριαρχία ενός κυρίως ατόμου και επιρροή ενός και μόνο στο κράτος. Σε ό,τι αφορά την νόμιμη παρουσία της, ε, της ΥΠΑ αρμοστίας του, ε, του ΟΗΕ, αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό. Γιατί αποστολή της ΥΠΑ της αρμοστίας και η μόνιμη παρουσία της εκεί είναι το καλύτερο εχέγγυο για τη διαφύλαξη των ε, προσφύγων. Και η πρόσφυγη είναι σημαντικό τμήμα των μεταναστών. Οι πρόσωποι της ΥΠΑ της αρμοστίας, παρόλο που δεν είχαν επίσημα άδεια μόνιμης παραμονής ήταν παρούσα στη Λιβύη για πολύ καιρό. Τώρα έχει συμφωνήσει να υπογράψει ε, και η Λιβύη αυτή την μόνιμη παρουσία της ΥΠΑ της Αρμοστής, να δεχθεί αυτή την παρουσία και μάλιστα να την εφοδιάσει με νομικό καθεστώς. Συνεχίζονται ε, μάλλον θα αρχίσουν εντό λίγο οι διαπραγματεύσεις Λιβύης και η της για τους πρόσφυγες. Δεν έχουν αρχίσει όμως ακόμη, αλλά αυτό το σημείο πραγματικά είναι κρίσιμο. Και εμείς με τις αρχές και τις ιδέες μας δεν μπορούμε να ε, εγκρίνουμε μια συμφωνία πλαίσιο αν δεν θεσμοθετηθεί και νομοποιηθεί η παρουσία της ΥΠΑ της αρμοστίας στη Λιβύη. Η Λιβύη έχει προσυπογράψει και τη σύμβαση του ΟΗΕ για την προστασία των προσφύγων, οπότε είναι λογικό να συνεργαστεί με την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία για την προστασία των προσφύγων. Υπάρχουν και άλλα αιτήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για παράδειγμα. Μπορούμε να τα υποβάλουμε χωρίς όμως να έχουμε την ψευδέστηση ότι θα γίνουν δεκτά ανεφόρων ή θα εφαρμοστούν αμέσως, αλλά τουλάχιστον θα δώσουμε κάποια ανάβσματα, θα, κάποια πίεση για τη μεταρρύθμιση. Άλλωστε υπάρχουν και εσωτερικές δυνάμεις, επιχειρηματίες που αντιλαμβάνονται την ανάγκη αυτών των μεταρρυθμίσεων στη Λιβύα. Οπότε ο ρόλος μας είναι να προωθήσουμε τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις. Γνωρίζουμε βέβαια ότι για τη Λιβύη πολύ σημαντικό είναι το, το σύστημα των θεωρήσεων. Τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ένωσης δεν είναι πρόθυμα να τροποποιήσουν το σύστημα θεωρήσεων, που είναι πολύ αυστηρό, αλλά μπορεί να βελτιωθεί, τουλάχιστον ως προς την προθεσμία για την παροχή θεώρησης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τέλος, η Λιβύη πέρασε από μια πολύ καχύπαπτη τακτική και θέση επένδυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξελίχθηκε λόγω της εκτίμησης που έδειξαν για το σχέδιο δράσης Μπενγκάζη με πρόταση της ε, Επιτρόπου Φέρερ Βάλτερ όταν κατάφερε να απελευθερωθούν οι πέντε νοσηλεύτερες από τη Βουλγαρία και ο Παλαιστίνιος γιατρός. Επίσης βοηθήσαμε τη Λιβύη να αντιμετωπίσει καλύτερα τα, θέματα, τα θύματα του AIDS. Με το σχέδιο αυτό εργασία είχαμε πολύ θετικά αποτελέσματα και η Λιβύη εκτίμησε ιδιαίτερε προσπάθειε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό άλλαξε την καχύποπτη αρχικά στάση που είχε απέναντί μα. Και μάλιστα αυτή η συνεργασία πια επεκτάθηκε και σε άλλε μεταδοτικέ ασθένειε, η βοήθεια τη προ τη Λιβύη. Αυτά δεν θα επεκταθώ άλλο γιατί έχετε λάβει το σχέδιο σύσταση. Παραλαμβάνω, η λύση δεν είναι να γυρίσουμε την πλάτη στη Λιβύη. Η Λιβύη είναι μια χώρα όπου το 1 τέταρτο του πληθυσμού της είναι αλλοδαπή ή μετανάστες εργαζόμενοι. Επίσης ε, ισχύουν πολλές διακριτικές ε, ε, πολλές διακρίσεις εις βάρος των μεταναστών αυτών. Μάλιστα στα αραβικά στη... ο όρος για τους μετανάστες είναι ε, ήλωτες. Και αυτό λέει πολλά. Είναι ελεηνή κατάσταση των μεταναστών, των εργαζομένων στη Λιβύη. Θα πρέπει λοιπόν ε, να κρατήσουμε αμύωτη την πίεσή μας και υψηλέ τις ε, απαιτήσει μας και υπό αυτό το πνεύμα συνέταξα και το σχέδιο έκθεσης, το σχέδιο σύστασης μάλλον. Ευχαριστώ. Στι 5 και 4 θα πρέπει να διακόψουμε την τακτική συνεδρίαση γιατί έχουμε μια συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών. Τέσσερις ομιλητέ έχουν ζητήσει το λόγο, αλλά παρακαλώ να είστε σύντομοι. Το λόγο έχει πρώτο ο κύριο Παντζέρη. Πάρα πολύ σύντομα. Θα συμφωνήσω με αυτά τα οποία έλεγε η Άννα Γκόμες έχει σημασία να είμαστε διατεθειμένοι σχετικά με τη Λιβύη να επιμείνουμε σε τρεις βασικούς τομείς. Είναι ένα συνομιλητής, τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε κατά προτεραιότητα και για θέματα τρομοκρατίας, ενέργειας, μετανάστευσης, ασφάλειας και στο τομέα της υγιεινής θα έλεγα. Και το κοινοβούλιο μας μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο ιδιαίτερα μετά από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης, της καινούργιας συνθήκης, που μπορεί να βοηθήσει στα πλαίσια της πολιτικής συνεργασίας. Δεν πρέπει να υποχωρούμε πάντα σε αυτά που απαιτεί ο Καντάφη, αλλά θα ήταν, θα έλεγα, λάθος να αγνοήσουμε την εκρηκτική κατάσταση την οποία αντιπροσωπεύει σήμερα η Λιβύη. Νομίζω ότι τα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση είναι αυτονόητα. Απαιτείται να υπάρξουν περαιτέρω βήματα σχετικά με την εφαρμογή της συνθήκης της Γενέβης και το άνοιγμα των γραφείων της ΥΠΑ της Θαυμοστίας. Δύο θέματα πρέπει να υπογραμμίσω επιπλέον. Είναι αλήθεια ότι εμείς έχουμε να κάνουμε με ένα δικτατορικό καθεστώς. Όμως, στα πλαίσια της σύστασης δεν πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό γιατί θυμάμαι ότι θα αυτοακυρωθούμε. Θα πρέπει να βρούμε μια διατύπωση έτσι ώστε αυτή η χώρα η οποία δεν έχει ιδιαίτερα δημοκρατικές τάσεις να εκπροσωπηθεί. Ένα δεύτερο θέμα πρέπει να, να επιμείνουμε περισσότερο. Υπάρχει ένα σημαντικό κέντρο το οποίο λειτουργεί αλλά είναι σχετικά περιορισμένο. Έχουμε τεράστιες παρουσίες ασθενειών μεταδοτικών και οι φορείς είναι πολλές φορές μετανάστες. Και αυτοί οι μετανάστες μπορεί να έλθουν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο πολύ εύκολα Συνεπώς το θέμα της υγιεινής πρέπει να τεθεί κατά προτεραιότητα στις συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά. Ε, Ευχαριστώ. Κύριος Κασουλίδης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γκόμες για την προσπάθεια που έκανε και τη σύσταση που συνέταξε. Τις περισσότερες φορές συμφωνώ μαζί της και σήμερα συμφωνώ με αυτό που είπε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τις επαφές με την Λιβύη, ότι υπάρχει θέμα ενεργειακής ασφάλειας, να επιμείνουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, παρουσία της υπατησαρμοστίας, αναστολή θανατικής ποινής κτλ. Διαφωνώ όμως κάθετα στο θέμα της ε, σύστασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διακόψει τι διαπραγματεύσει για τη Συμφωνία Επανειστοχής και να την αποσυνδέσει από τη Γενική Συμφωνία Πλαίσιο που διαπραγματεύεται με τη Λιβύη. Καταρχήν κύριε Πρόεδρε, δεν καταλαβαίνω το λόγο αυτής της πρότασης. Ήταν κατεπήγον να επισέλθουμε στο θέμα αυτό με τη συνοπτική διαδικασία, με ταχεία διαδικασία, το fast track. Και σίγουρα η διαπραγματευτική φάση του Ιανουαρίου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα είναι η τελευταία. Θα έχουμε πολλές διαπραγματευτικές συναντήσεις. Και δεδομένων των δυσχερών πτυχών και των δυσκολιών αυτών των συμφωνιών, προτάθηκε να αποσυνδεθεί το θέμα της συμφωνίας πλαισίου από την συμφωνία επανεισδοχής. Παρ' όλα αυτά, η Λιβύη θα εφαρμόσει ε, επανεισδοχή για τους δικούς της υπηκόους και αρνείται κατηγορηματικά να αναλάβει ευθύνη για τους υπηκόους των τρίτων χωρών, όπως και άλλες μεσογειακές χώρες. Η Επιτροπή δεν ε, είναι αισιόδοξη για τη μεταστροφή της Λιβύης, αλλά ίσως αυτό συμβεί αργότερα, γιατί πάντα τα επίμαχα θέματα μένουν για το τέλος της διαπραγματεύσης. Οπότε εδώ δεν έχουμε να κάνουμε τόσο με την απόρριψη, με την άρνηση της Λιβύης να συζητήσει θέματα των χωρών, αλλά έχουμε και το Μαρακό και άλλες μεσογειακές χώρες, τρίτες χώρες, που διαμαρτύρονται γιατί δόθηκαν ε, ε, καθεστώτα διευκόλυνση θεωρήσεων με τις χώρες ε, της Ανατολικής Γειτονίας, κάτι που θεωρούν διακριτική μεταχείριση εις βάρος των χωρών ε, γειτονίες ε, με τον Νότο, κυρίως ε, των γειτονικών χωρών της Μεσογειακής Λεκάνης. Βέβαια, διευκόλυνση στις θεωρήσεις δεν σημαίνει κατάργηση θεωρήσεων. Απλώς δίνεται πιο σύντομα η θεώρηση ή θέματα κατηγοριοποίησης θα μπορούσαν να εξεταστούν από το Συμβούλιο. Μάλιστα το Συμβούλιο θεώρησε τη Λιβύη ως σημαντική πύλη εισόδου των μεταναστών προς την Ευρώπη. Το ίδιο, το ίδιο ίσχυσε για την Τουρκία. Και μάλιστα στη διάσκεψη κορυφή του Ιουνίου αναφέρθηκαν ρητά αυτέ οι δύο χώρε, Τουρκία και Λιβύη. Οπότε δεν είναι ότι ε, επειδή η Τουρκία δεν έχει συμφωνία επανεισδοχή, το ίδιο θα πρέπει να αποφευθεί και με τη Λιβύη. Δεν είναι επιχείρημα αυτό. Το πρώτο μα μέλημα θα πρέπει να είναι η Μάλτα. Γιατί η Μάλτα είναι η χώρα που δέχεται το πρώτο κύμα των λαθρομεταναστών. Και είναι μικρή χώρα. Όχι μόνο δεν μπορεί να αντέξει αυτό το μεταναστευτικό ρεύμα, αλλά υπάρχει και δημογραφικό ζήτημα. Μετά έχουμε την Ιταλία. Η Ιταλία συνήψε το 2008 μια συμφωνία φιλίας που οδήγησε στη μείωση ε, αποστολής λαθρομεταναστών από τη Λιβύα προς την Ευρώπη από τη Λιβύη προς την Ευρώπη. Αυτό όμως δεν ανταποκρίνεται στις δικές μας ανησυχίες για την εφαρμόγη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το να ζητούμε λοιπόν τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διακόψει τι διαπραγματεύσει για τι συμφωνίε επανειστοχή, όχι μόνο θα αποδυναμώσει η διαπραγματευτική ικανότητα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα δώσουμε και κακά παραδείγματα προ άλλε χώρε τη Μεσογειακή Λεκάνη, τρίτε χώρε με τι οποίε συζητούμε θέματα επανειστοχή. Πιστεύω ότι αυτά τα θέματα θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με γενικότερο τρόπο στα πλαίσια τη Ένωση για τη Μεσόγειο. Και αυτή η διαπίστωση και η διάγνωση είχε γίνει από την αρχή να συνάψουμε συμφωνίες επανιστοχής σε ολόκληρη τη Μεσογειακή περιοχή. Και όταν μιλούμε για επανιστοχή δεν εννοούμε ούτε τούντες άσυλο, ούτε πρόσφυγες, ούτε άτομα χρήζοντα προστασίας. Μιλούμε για λάθρομετανάστες. και όταν υπάρχει κίνδυνος είτε βασανιστήριων, είτε απάνθρωπης ε, μεταχείρισης, είτε θανατικής ποινή, μπορούμε ε, να ενισχύσουμε την προστασία στα πλαίσια του δικαιώματος ε, μη επαναπροώθησης. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Φλότ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, γιατί μας αφήσετε πολύ ελεύθερο στο χρόνο. Ελπίζω αυτό να ισχύσει για όλους αυτή η επίοικια ως προς τη διαχείριση του χρόνου. Ευχαριστώ την Αναγκόμες για την σύστασή της, για την έκθεσή της. Βέβαια θα ήταν πολύ πιο εύκολο για μας να επικεντρωθούμε στα κέρια σημεία της διαπραγματευτικής εντολής, αλλά δεν γνωρίζουμε το ακριβές περιεχόμενο αυτής της εντολής, δυστυχώς. Και έτσι το Συμβούλιο δεν τηρεί τι υποχρεώσει που έχει με βάση τη νέα συνθήκη τη Λισαβόνα. Και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε από την αρχή, γιατί πρέπει ήδη να είχαμε λάβει την εντολή για του όρου τη εντολή. Θα ήθελα να σχολιάσω δύο παρατηρήσεις των προλαλισσάντων, Παντζέρη και Κασουλίδη. Ίσως ε, έγινε κάποια παρεξήγηση. Δεν φαντάζομαι να διανοείται κανείς ότι οι ε, μετανάστες είναι αυτοί που μεταφέρουν τις μεταδοτικές ασθένειες στην Λιβύη, γιατί και οι νοσηλεύτες από τη Βουλγαρία ήταν ε, μετανάστερες. Αυτό μάλιστα έλεγα τότε όταν είχα πάει και εγώ στη Λιβύη, πρόσφατα σχετικά το 2005 και από τότε το άκουγα, ότι οι μετανάστες και είναι πολύ άριθμοι γιατί ε, στα 5 εκατομμύρια κατοίκους, στα 2 εκατομμύρια είναι μετανάστες. Είναι πραγματικά τεράστια η αναλογία. Αδιανόητο για μας στην Ευρώπη. Έλεγαν τότε ότι οι μετανάστες είναι οι φορείς των ε, νόσων και μάλιστα 80% των... και ήταν, ε, ήταν ε, ένοχοι για το 80% των εγκλημάτων. Αυτά έλεγαν τότε οι, Λιβύοι, οι αρχές της Λιβύης. Δεν λαμβάνουμε φυσικά υπόψη σοβαρές τέτοιου είδους καταγγελίες αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων. Ίσως θα πρέπει να αναλάβουμε πιο συγκεκριμένα επιχειρήματα εδώ, γιατί ο ρατσισμός κατά το μαύρο στη Λιβύη είναι πραγματικά βάναυσος. Θα πρέπει να το πούμε πιο ρητά ίσως το κείμενο. Και αυτά λένε και στη Λιβύη κύριε Κασουλίδη, ότι δεν έχουν πρόβλημα ασύλου και ε, διεθνούς προστασίας, γιατί τα δύο εκατομμύρια μεταναστών είναι οικονομικοί μετανάστες και έρχονται για να βρουν δουλειά στη Λιβύη. Κι όμως έχουμε πολλές ε, περιπτώσεις, οι πρόσφατα με κατοίκους Ερυθρέας, που δείχνουν ότι πολλοί μετανάστες που θέλουμε να εργαστούν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας, θα πρέπει να δίνονται να έχουν πρόσβαση σε σαφή διαδικασία και το γραφείο της ΥΠΑ ε, αρμοστίας είναι το ελάχιστο, ούτε καν είναι το εχέγγυο μιας ε, θεμητής διοικητικής ε, ή κρατικής διαδικασίας για πρόσβαση σε αίτηση ή πρόσβαση σε άσυλο μάλλον. Θα πρέπει αυτό να το πούμε σαφώς στο κείμενο. Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε και γι' αυτό θα συντάξουμε και τροπολογίες είναι να παρακολουθήσουμε αυτό το διάλογο, να στηρίξουμε όλες τις προσπάθειες που έχουν στόχο την γενικότερη βελτίωση της κατάστασης, ώστε να γίνει πραγματικότητα ο σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου στη Λιβύη, γιατί όπως είπε και η κυρία Γκόμες, η Λιβύη είναι δικτατορικό καθεστώς. Και όταν λέμε δικτατορία, εννοούμε ότι υπάρχει τεράστια δυσκολία ε, να βρεθούν ανεξάρτητες οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, στους οποίε μπορούμε να στηριχθούμε, προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση της συνεργασίας που έχουμε με τις αρμόδιες αρχές. Θα το συζητήσουμε αύριο και στις συνεδρίες των σχεδόν εισηγητών, αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε πιο συγκεκριμένες προσπάσεις. Πέρα την ανάγκη ενθάρρυνσης, ε, προσπάθειας να πείσουμε τη Λιβύη και τα λοιπά και πίεσης, χρειάζονται και κάποια πιο συγκεκριμένα σημεία, αν θέλουμε νυφάλια να εξετάσουμε μια συνεργασία με τη χώρα αυτή. Η ε, κυρία Ότζελαν. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, συμφωνώ ότι είναι πολύ καλή αυτή η έκθεση, το σχέδιο τουλάχιστον. Δεν θα επαναλάβω τα σχόλια των συναδέλφων. Θα συντάξω και κάποιες τροπολογίες. Και εγώ είχα εμπειρία διαβίωσης υπό δικτατορικό ζυγό ή σε αυταρχικό καθεστώς και αντιλαμβάνομαι πόσο δύσκολο είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει σχέση με μια χώρα σαν τη Λιβύη. Αυτό είναι βέβαια ένα το κρατούμενο, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά το θέμα της, του γραφείου μας στην Τρίπολη. Αυτό σημαίνει θα έχουμε στενότερες σχέσεις και θα μπορέσουμε να επηρεάσουμε περισσότερο εμείς ως κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία τις σχέσεις αυτές με τη Λιβύη. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ζητήσουμε την ε, ίδρυση ενός ε, γραφείου στη Λιβύη, στην Τρίπολη. Αλλά σημαντικό θα ήταν και η Λιβύη να εκδηλώσει προθυμία συνεργασία και ανάπτυξη ή σύσφυξη των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να συμμετέχει στι δραστηριότητε τη Ένωση για τη Μεσόγειο. Και αυτό θα πρέπει να το δηλώσουμε πιο ρητά. Και αυτό το θέμα τη αναστολή των θανατικών καταδικών ή άλλα ζητήματα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να τα τονίσουμε όλα αυτά ίσως με πιο κατηγορηματικό τρόπο από ό,τι αναφέρονται μέχρι στιγμή στο σχέδιο έκθεσης. Ευχαριστώ κυρία Ογιουλάντ ιδιαίτερα που τηρήσατε το χρόνο σας. Παρακαλώ το ίδιο να κάνουν και οι δύο τελευταίοι ομιλητές, ο κύριος Μάουρο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ θερμά την κυρία Γκόμες που τόνισε δύο πολύ σημαντικές πτυχές. Το πρώτο είναι ο βασικός στόχος. Ξαναρχίζει ο κύριος Μαύρος συγχαίροντας την κυρία Γκόμες. Δύο πλευρές να υπογραμμίσω. Η πρώτη σχετική με το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να αναπληρώσει μια, ένα κενό θα έλεγα το οποίο καλύπτεται από διμερείς εθνικές συμφωνίες. Η δική μου χώρα θα έλεγα υπόκειται σε μια συμφωνία η οποία κανονικά θα έπρεπε να είχε γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παλιά λέγαμε ότι η Μάλτα από μόνη της τόσο μικρή δεν μπορεί να επιβραδύνει το μεταναστευτικό φαινόμενο αλλά και η Ιταλία δεν μπορεί σε ένα θέμα τόσο περίπλοκο και σύνθετο να αναλάβει τις ευθύνες όλων. Και γι' αυτό να περιγράψω λίγο τις τροπολογίες οι οποίες θα κατατεθούν από πλευράς μου. Θα κατατεθούν γιατί κάποια από τα θέματα που έχουμε μπροστά μας μας δείχνουν τη μοναδικότητα της περίπτωσης της Λιβύης. Είναι αλήθεια ότι η Ιταλία έχει υπογράψει μια κάποια συμφωνία πρόσφατα, το 2008, και δεν μπορούν φυσικά να εφαρμοστούν μέσα σε ένα μήνα από μια άλλη κυβέρνηση. Αλλά είναι μια συμφωνία η οποία προσπάθησε η, ελληνική, η Ιταλική κυβέρνηση για δεκαετίες να προετοιμάσει, ακριβώς γιατί ήταν απούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και απόν είναι και ο ΙΕ έχει βάλει πρόεδρο Λίβιο ε, στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΙΕ. Μήπως θα έπρεπε να επιβάλλει και την παρουσία του εκεί ε, στα πλαίσια της ε, ΥΠΑ της Αρμοστίας. Ελπίζω οι τροπολογίες μου να γίνουν δεκτές από την εισηγήτρια. Ευχαριστώ κύριε Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ. Δύο σχόλια έχω. Ένα επί της ουσίας και ένα επί της διαδικασίας. Ως προ την ουσία, ευχαριστώ την κυρία Γκόμες για το εξαιρετικό έργο που έχει πραγματοποιήσει αυτό το σχέδιο ψηφίσματος. Άλλωστε μας έχει συνηθίσει σε πολύ αξιόλογες προσπάθειες. Είναι πραγματικά ιδιάζουσα η κατάσταση με μια ιδιαίτερη χώρα που χαίρει και ειδικού καθεστώτο. Θα ήθελα να πω ότι ω προ την ουσία ο αντιπρόεδρος της ομάδας μας, ο κ. Κασουλίδης, εξήγησε την ε, επίσημη θέση του ΕΛΚ και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που μας είπε ο κ. Κασουλίδης. Κυρία Γκόμες, σε ό,τι αφορά την αναστολή διακοπή των ε, συμφωνιών επανεισδοχής, αυτό είναι πολύ λεπτό ζήτημα και όπως είπε ο κύριος ε, Μάουρο, χώρες όπως η Μάλτη υφίσταται τεράστια μεταναστευτική πίεση. Πολλοί επίτροποι πραγματοποίησαν επισκέψεις στη χώρα. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια πολιτική που δεν θα εφαρμόζει διακρίσεις εις βάρος της χώρας, αλλά όπως είπε και ο κύριος Παντσέρη, αν θέλουμε μια realpolitik, θα πρέπει να πάρουμε τον παλμό της κατάστασης και να προσέξουμε στη διατύπωση του κειμένου. Αλλά θα μπορούσαμε, κυρία Γκόμες, να βρούμε μια διατύπωση, ώστε να συνδυάσουμε και τις προσπάθειες για σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με τη λογική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προωθήσει τη Συμφωνία Επανιστοχής. Γιατί στην Ευρώπη πολλές ε, γειτονικές χώρες της ε, Λιβύης είναι πιθανά θύματα μιας αποτυχίας τέτοιων συμφωνιών. Κυρία Γκόμες, γνωρίζετε ότι τρέφω ιδιαίτερη ιστορία απέναντί σας και έχω ιδιαίτερη εκτίμηση προς το έργο σας, αλλά Επαναλαμβάνω, ο κέντρο μα ηγητή είναι ο κύριο Κασουλίδη. Σα με διορθώσει αν κάνω λάθο, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σύντομη η διορία για τι ε, τροπολογίε. Γιατί αν δεν κάνω λάθο, ε, σήμερα στι 5 το βράδυ μα λέτε ότι ε, λίγη προθεσμία αύριο το μεσημέρι. Εγώ δεν πρόκειται να καταθέσω τροπολογίε, αλλά δεν ξέρω αν ε, οι σκιώδει ηγητέ είναι ικανοποιημένοι με αυτή την πολύ βραχία προθεσμία για τι τροπολογίε. Αυτά κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε κυρία Γκόμες και συμφωνώ απόλυτα με τη θέση που εξέφρασε ο σκιώδης μας ηγετής ο κύριος Κασουλίδης. Θα ήθελα να επιθυμίσω ότι η διορία για τις τροπολογίες λήγει στις 2 Δεκεμβρίου. Η κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις. Συμφωνώ, συμφωνώ ότι το σημαντικότερο πρόσκομα είναι το θέμα της εμφανίας της επανεισδοχής. Θα το συζητήσουμε και αυτό και άλλα θέματα στη συνάντηση που θα πραγματοποιήσουμε αύριο με τους σκιώδεις συγητές. Τώρα γιατί είναι τόσο βραχή αυτή η διορία για τις, τροπολογίε. για τροπολογίες. Μην ξεχνάτε ότι αυτό είναι ένα σχέδιο έκθεσης, ε, σχέδιο σύστασης, γιατί περιμένουμε ακόμη το, τη συμφωνία πλαίσιο, το σχέδιο συμφωνίας πλαίσιο. Εμείς προσπαθούμε να επηρεάσουμε την τελευταία φάση των διαπραγματεύσεων που θα λάβει χώρα τον Ιανουάριο. Γι' αυτό ζητήσαμε κάπως εσπευσμένη διαδικασία, ώστε να εθετήσουμε την έκθεση στην Ολομέλεια του Ιανουαρίου. Βέβαια, από εσάς εξαρτάται, επαφίεμαι στα χέρια των συναδέλφων και των ομάδων. Εγώ κάνω τη δουλειά μου, είμαι εδώ πρόθυμη για να το διαπραγματευτώ με τις πολιτικές ομάδες. Αν δεν προλαβαίνουμε για τις αρχές Ιανουαρίου, εντάξει, πάντως δεν νομίζω ότι η Επιτροπή θα ολοκληρώσει τη διαπραγματεύση μέχρι τέλη Ιανουαρίου. Να δούμε τι θα μας πει και η Επιτροπή. Πάντως το γεγονό ότι ήδη συζητούμε το θέμα και ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις σημαίνει ότι μπορεί να αρχίσει και η επιρροή μας στην πορεία των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Bon, donc délai des amendements. Καλώς, οπότε η προθεσμία για τις τροπολογίες λήγει στις 2 Δεκεμβρίου για να εγκρίνουμε την έκθεση 9 Δεκεμβρίου εκτός και αν για πολιτικούς λόγους ε, μετατοπιστεί αυτή η διορία. Ωραία, λύεται η τακτική συνεδρίαση. Σε λίγο θα αρχίσει η συνεδρίαση και κλεισμένο των θυρών. Οπότε όσοι δεν δικαιούνται να παραμείνουν στην αίθουσα παρακαλώ να την εγκαταλείψουν.